Werte κυρίε και κύριοι, επεξηγήσει ψήφων. Έκθεση Σικέσκη. Καταρχά, ποσοστό αναπροσαρμογή για τι άμεσε ενισχύσει αφορά το 2015. Ο κύριο Πέτερ Γιάρ. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Και καλώ του λοιπόν συναδέλφου, εφόσον δεν θέλουν να παραμένουν να αποχωρήσουν από την αίθουσα ώστε να μπορέσουν όσοι έχουν να κάνουν επεξήγηση ψήφου να μιλήσουν. Κύριε Γιάος, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Γιατί, ναι, πολύ ωραία το λένε ότι είναι μια